Shall we start, ladies and gentlemen? Να ξεκινήσουμε. Σας καλωσορίζω κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι. Στην ενδιαφέρουσα αυτή συνάντηση, συνεδρίαση, που το μοναδικό της πρόβλημα είναι ότι διεξάγεται πέμπτη απόγευμα και βλέπετε ότι οι συναδελφοί έχουν πάρα πολλή δουλειά και γι' αυτό θα είμαστε Θα είμαστε πιο μοναχικοί σήμερα το απόγευμα. Έχουμε όμως ε, ενδιαφέροντα θέματα. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μαύρη Θάλασσα είναι η πρώτη μας ε, γνωμοδότηση με εισηγήτρια την κυρία Τικάου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Πρόκειται για την ανάγκη Μιλάμε για την ε, ανάγκη πιο αντιμετωπίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Μετά την τελευταία διεύρυνση κατέστη σημαντικό παράγοντα η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περιοχή αυτή και μάλιστα με ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία για την διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δεδομένη τη εγκύτητά τη με την Κασπία Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία. Στην ε, γνωμοδότησή μου αναφέρομαι στη μακρόχρονη στρατηγική τελική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωσης και Ρωσία και τα κοινά συμφέροντά τους σε ό,τι αφορά την προώθηση του διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων στην περιοχή. καθώς και στη διευκόλυνση και την ελευθέρωση του εμπορίου στην ε, περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Μιλώ επίσης για νέες διασυνδέσεις φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Και μιλάμε για σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε πάσης φύσεως. Και επίσης θα πρέπει να γίνουν νέες επενδύσεις στην περιοχή. Και να υπάρξουν και ίσες, ε, ε ίσοι όροι για τις επενδύσεις στην περιοχή σε ό,τι αφορά την πολιτική ασφάλεια ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή βασίζεται στην διαφοροποίηση των πηγών και εδώ θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του αγωγού φυσικού αερίου Ναμπούκο και επίσης την έκθεση από αυτήν την έκκληση προς την Επιτροπή να επιταχύνει την υλοποίησή του σχεδίου του Ναμπούκο. Περαιτέρω σχέδια περιλαμβάνουν την, ε, το δίκτυο μεταξύ Τριέστης και Κωνσταντσάς... για το πετρέλαιο. Και αναφέρεται και η διασφάλιση του αγωγού από την Γεωργία προς την Κωνσταντσά. Θα ήθελα να τονίσω με την γνωμοδότηση αυτή ότι τα ενεργειακά δίκτυα πρέπει να λειτουργούν με αμφίδρομο τρόπο. Σε ό,τι αφορά θέματα έρευνας, θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικά προγράμματα. Αναφέρω ενδεικτικά το Interconnection και το Black Sea Πρόκειται για ένα περιφερειακό δικτύο και καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την πρόθεση των ε, ερευνητικών προγραμμάτων στην περιοχή όπως το SIN, το GRID, το HPC και το καθεξής. Να αναφέρω επίσης περαιτέρω ότι είναι απαραίτητο σε ό,τι αφορά να βελτιωθούν οι υπηρεσίε ε, στους λιμένες, σε ό,τι αφορά την προμήθεια πετρελαίου και αερίου. Και να διασφαλιστεί επίσης η διαλειτουργικότητα των φορέων, προκειμένου να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των μεταφορών στη θάλασσα και μέσω ξηράς. Δυστυχώς, ως τώρα, ο εύξηνος πόντος αποτελούσε τη μοναδική θάλασσα για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε ακόμα επενδύσει σε ό,τι αφορά τις πλωτές οδούς. Ελπίζω να διατεθούν κονδύλια από το TNT, από τα διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών. Επίσης, η συνεργασία σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα στη Μαύρη Θάλασσα θα πρέπει να λάβει μια όθηση. Όλα αυτά φυσικά βάσει της νομοθεσίας αναφορικά με την ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζουμε επίσης την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των χωρών της Μαύρης Θάλασσας με τη συμπερίληψη και των κατάλληλων χρηματοοικονομικών μέσων. Δεδομένη της ε, σημασίας της Επιτροπής Ευξήνου Πόντου και της ε, σημασίας της περιοχής, καθώς και τη σημασία του έργου που διεξάγεται από όλους τους παράγοντες, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταστεί πιο δραστήρια στον τομέα αυτό, Γι' αυτό καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μια στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα, η οποία θα πρέπει να υποστηριχθεί και από ένα σχέδιο δράση στου παρακάτω τομείς συνεργασίας, αηφόρο οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση των συστημάτων διασύνδεση και επικοινωνία, πρόσταση του περιβάλλοντο, ασφάλεια, μετανάστευση και πολιτιστικέ αλλαγέ, χρησιμοποιώντα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα. Και εδώ να τονίσω και να υπογραμμίσω ότι υπάρχει ένα λάθος ε, στην ρουμανική μετάφραση στα αγγλικά αναφέρεται flagship project, στρατηγικά project. Στα ρουμανικά μεταφράστηκε ως πιλωτικά προγράμματα. Ο όρος αυτός θα υποβάλω διορθωτικό, γιατί μιλάμε για στρατηγικά σχέδια για τον εύξονο πόντο και γι' αυτό Θα πρέπει να γίνει αυτή η διόρθωση. Επίσης να προσθέσω ότι το σχέδιο δράσης που θα πρέπει να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι εύκολο στη σύνταξή του, στην κατάρτισή του, γιατί υπάρχουν ήδη τρεις εταιρικές σχέσεις σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συνέργειας ε, για τον εύξηνο πόντο μιλάμε για το περιβάλλον, τις μεταφορές, ε, για αυτές είναι υπεύθυνη η Ελλάδα και επίσης για την ενέργεια. Για την ενέργεια υπεύθυνη είναι η Βουλγαρία. Αυτές ε, οι εταιρικέ σχέσεις αφορούν και κάποιες ε, δράσεις στην περιοχή, αλλά και τη γενικότερη στρατηγική στην περιοχή. Χρειάζεται όμως ένα ευρύτερο πλαίσιο, μια γενικότερη στρατηγική, πέρα από τις μεμονωμένε τράσεις και τις μεμονωμένε τομείς. Ελπίζω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταπεξέλθει σε αυτές τις νέες προκλήσεις στην περιοχή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, κυρία Τικάου, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Να ομολογήσω ότι μπορεί να είμαστε λίγοι στον αριθμό, αλλά Έμαθα σημαντικά πράγματα και σας ευχαριστώ γι' αυτό και ο συνάδελφος Μπίπαλ παίρνει πρώτος το λόγο. Ja, vielen äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Äh, e Από πλευράς ΕΛΚ πρέπει να πούμε ότι συμφωνούμε με την γνωμοδοτησία αυτή, η οποία παρέχει την βέλτιστη πλατφόρμα ως προς την στρατηγική για την αξιοποίηση του σημαντικού δυναμικού της περιοχής, για την ευφυή διασύνδεση e, των τομέων αυτών και για την εφαρμογή σημαντικών τομέων όπως είναι η ενέργεια. Η στρατηγική αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και η γνωμοδότησή σας θεωρώ ότι αναφέρεται με μοναδικό τρόπο στα θέματα ε, της ε, Μαύρης γιατί είναι η πρώτη φορά που διαβάζω ένα κείμενο που αναφέρεται στο στο συνδυασμό των υφιστάμενων μέσων πρέπει να ομολογήσω ότι ποτέ τα τελευταία έξι χρόνια δεν έχω δει να προτείνεται αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων μέσων, να μην προτείνεται επιπλέον χρηματοδότηση. Το μοναδικό που λείπει, θεωρώ, είναι η αναφορά στη στρατηγική του Δούναβη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει εγκύτητα και άρα υπάρχουν στρατηγικά πεδία τα οποία θα πρέπει να αναφερθούν. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα υποβάλλουμε Τροπολογίε. Ευχαριστούμε, λέει ο, ο πρόεδρος, τον κύριο Πίπερ. Ζητά κάνει άλλο το λόγο. Σω από θέλει κάποιος άλλος κοιότης συζητητής να πάρει το λόγο. Η κυρία Τσιμάσκη, αν δεν ζητά κανεί άλλο το λόγο, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει θέση. Δεν ξέρω αν παρευρίσκεται κανεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ich kann's nicht lesen. Entschuldigung. Μπορώ να διαβάσω το όνομά σας. Σας ζητώ συγγνώμη. Uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την ε, εμπεριστατωμένη της παρουσίαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με πολλά από τα σημεία που παρουσίασε η συγγήτρια. Θα ήθελα πάντως να υπογραμμίσω ότι πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή να εδραιώσουμε τη συνέργεια για τον εύξηνο πόντο, την πρωτοβουλία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του εύξηνου πόντου, που εγκαινιάστηκε το 2008 στην Υπουργική διάσκεψη του Κιέβου, στην οποία συμμετείχαν οι Υπουργοί ε, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Υπουργοί των χωρών ε, της Μαύρης Θάλασσας. Ακόμη δεν την έχουμε υλοποιήσει αυτή την πρωτοβουλία της συνέργειας για τον εύξενο πόντο. Αυτή την ε, πρωτοβουλία θα πρέπει πρώτα να εδραιώσουμε πριν περάσουμε σε άλλα βήματα. Αναφέρθηκαν οι τρεις εταιρικές σχέσεις στο περιβάλλον, τις μεταφορές και την ενέργεια. Στην πράξη όμως ε, μία μόνο εγκαινιάστηκε, η εταιρική σχέση για το περιβάλλον. Και αυτό φέτος. Οι άλλες δύο δρομολογούνται. Και αυτό δεν οφείλεται σε καμία κολλησιεργία ή οκνηρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε σε έλλειψη ενδιαφέροντος από τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε για να παραδεχτούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και το βασικό πρόβλημα είναι ότι κάποιες μεγάλες χώρες της περιοχής αισθάνονται δυσφορία με την προσπάθεια εντονότερης παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Γιατί Τώρα πια, εκτός από την Ελλάδα, έχουμε και δύο άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι παράκτιες της Μαύρης Θάλασσας, το Αυξηνοπόντο, όπως αναφέρθηκε η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας εκεί. Δεν, είμα, δεν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στη Βαλτική θάλασσα ή στην α, θάλασσα του Μπάρεντς. Υπάρχουν και άλλες γειτονικέ χώρες. Γειτονικέ όχι με την τεχνική έννοια τώρα, αλλά με τη γεωγραφική. Αυτή λοιπόν είναι η θέση μας. Εμείς πιστεύουμε ότι πρώτα θα πρέπει να εδραιώσουμε τη συνέργεια για τον εύξηνο πόντο, γιατί είναι καλή πρωτοβουλία και χρησιμοποιεί τα εργαλεία και τους μηχανισμούς που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει και την διαπεριφερειακή συνεργασία εντός ευρύτερης περιοχής, αλλά να προωθήσει και τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιοχής του εύξηνου πόντου. Βέβαια, Αντιλαμβάνομαι ότι οι αρμοδιότητες της Επιτροπής που είναι κυρίως η βιομηχανία σας υποχρεώνουν να στραφείτε κυρίως σε αυτή την πτυχή της στρατηγικής για τη Μαύρη Θάλασσα, τη βιομηχανική. Αλλά η συνεργασία στην περιοχή του εύξηνου πόντου δεν περιορίζεται στην ενέργεια. Παρόλο που η ενέργεια είναι κρίσιμος ε, και ναυραλγικός τομέας, αλλά προχωρούμε και σε άλλους τομείς, όπως είναι η διασυνοριακή συνεργασία. Και για πρώτη φορά στην ιστορία θα έλεγα, παρόλο που δεν θέλω να δραματοποιώ τα πράγματα, για πρώτη φορά λοιπόν έχουμε διασυνοριακή συνεργασία και διακρατική διασυνοριακή συνεργασία στην ε, Μαύρη Θάλασσα. Δεν είναι βέβαια τόσο φιλοδοξό όσο το αντίστοιχο της Βαλτικής, αλλά είναι το πρώτο τέτοιο βήμα. Δεν είχαμε προηγούμενο η πείρα στον τομέα αυτό προηγουμένως. Και είχαμε την περίοδο 2007-2013 που είναι η πρώτη περίοδος που γίνεται η αρχή αυτών των βημάτων και στην επόμενη περίοδο των δημοσιονομικών προοπτικών ελπίζω ότι θα χρηματοδοτήσουμε τα ψηλέστερα, τα πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα που έχουμε σε αυτή την περιοχή. Γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε βήματα προόδου και επιμένω εδώ στην πρόοδο για να βρούμε ε, λύση και να χαλαρώσουμε μερικές τεταμένες περιοχές. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Να δώσω το λόγο και πάλι στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ειλικρίνειά της σε ό,τι αφορά τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να εργάζεται προκειμένου να καταρτήσει μια στρατηγική για την ε, Μαύρη Θάλασσα. Διάβασα πρόσφατα ότι η Ρωσία θέλει να εξάγει αέριο προς την Ασία, προς την Κίνα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η εκείτητα του εύξηνου πόντου θα μπορούσε λόγω της εγκύτητας με την ε, Κασπία να τονώσει την ανεξαρτησία ως προς την ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποφύγει και δεν πρέπει να αποφύγει να καταστρώσει μια στρατηγική για τον εύξηνο πόντο. Και θα ήθελα να πω ότι στην περιοχή αυτή υπάρχει μια τεράστια δραστηριότητα βιομηχανική. Φυσικά, κάθε χώρα έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, αλλά θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε μια συνεργασία η οποία θα απέβαινε ε, επωφελής για όλα τα κράτη. Επιπλέον να αναφερθώ στο σημείο 8 της γνωμοδότησης της ΙΤΡΕ, της, της Επιτροπής Βιομηχανίας δεν περιοριζόμαστε στον τομέα της ενέργειας. Προτείνουμε και ένα σχέδιο δράσης με πρωτοποριακά προγράμματα σε πολλαπλούς τομείς, όπως ε, είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η βελτίωση της δικτύωσης και της επικοινωνίας. Όλα αυτά. Προστασία του περιβάλλοντος, μετανάστευση, πολιτιστικές ανταλλαγές. Είναι πολλαπλές ε, οι προτάσεις μας φυσικά και ο τομέας της ενέργειας είναι στρατηγική σημασία για την Ένωση. Αλλά αποτελεί ένα τμήμα μόνο των προσπαθειών που θα πρέπει να καταβληθούν στον τομέα του εύξηνου πόντου. Αυτό που θέλω να υποστηρίξω το εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη σημασία στην περιοχή αυτή. Και αυτό θα επιτευχθεί με μια στρατηγική στην ε, περιοχή, με βάση φυσικά την ισότητα όλων των εμπλεκομένων φορέων. Φυσικά με χαρά θα ακούσω και τις θέσεις των συναδέλφων, αλλά είμαι απόλυτα αποπισμένη, όπως είπα και προηγουμένως, ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική πολιτική του της Ένωσης και να προσπίσει τη θέση του. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, να σας πω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι στις 12 η ώρα στις 12 Οκτωβρίου και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το 17. ΑΕΠ, η μέτρηση της προόδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Η συνάδελφος Ματίας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δηλώσω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι συζητάμε αυτό το θέμα και ότι προσπαθούμε να λάβουμε θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Όλοι γνωρίζουμε ότι το ΑΕΠ ως όργανο μέτρησης και αξιολόγησης της επιτυχίας των οικονομικών πολιτικών είναι περιορισμένο. Έχει αποδειχθεί αυτό. Και επίσης συνδέεται περισσότερο με την παραγωγή και ελάχιστα με την ευημερία και το βιωτικό επίπεδο. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό της ανεπάρκειας του έπος μέτρου ε, ως οργάνου μέτρησης. Θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε και κάποιους ε, συμπληρωματικούς δείκτες πέραν από αυτών που υπάρχουν ήδη και ως θεμελιώδη στόχο μας να έχουμε τη συγκέντρωση διεξοδικών ε, πληροφοριών που θα αποτελέσουν τη βάση για τη χάραξη των πολιτικών. Επαναλαμβάνω, το ΕΠ είναι ένα όργανο μέτρησης που συνδέεται κυρίως με την παραγωγή δεν εκπροσωπεί σωστά την αξιολόγηση των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών. Ω εκ τούτου θα πρέπει να θεσπιστούν, επαναλαμβάνω, συμπληρωματικοί δείκτες που θα πρέπει να περιλαμβάνουν κοινωνική διάσταση, περιβαλλοντική, αναπτυξιακή, βιωτικού επίπεδου, έρευνας, ε, επίπεδου απασχόληση Θα μπορούσαμε να συντάξουμε ένα πιο εξαντλητικό κατάλογο, αλλά δεν χρειάζεται. Ενδεικτικά τέτοιου είδους δείκτες θα έπρεπε να, να θεσπιστούν συμπληρωματικά. Επίσης, πιστεύω ότι οι συμπληρωματικοί δείκτες ε, του ΑΕΠ θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη μακροοικονομική δραστηριότητα, κάτι που δεν γίνεται επαρκώς σήμερα. Έτσι θα πρέπει να παρελάβουμε και μη εμπορικές πτυχές στον υπολογισμό και θα πρέπει να ληφθούν και θετικοί εξωτερικοί παράγοντες και αρνητικοί εξωτερικοί παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας, για, όπως είναι η εγχώρια παραγωγή ή άλλοι διαστάσεις που αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνονται υπόψη. Και επίσης ε, θα ήθελα να πω το εξής. Σε ό,τι αφορά το έργο της Επιτροπής, είναι σημαντικό ότι για να υλοποιήσουμε τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αν κρατήσουμε το ΑΕΠ ως ε, μοναδικό όργανο μέτρησης και δεν το συμπληρώσουμε με άλλους δείκτες, αναγκαστικά το ΑΕΠ θα μειωθεί. Οπότε οι νέοι δείκτες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να αξιοποιούν όλα αυτά τα στοιχεία. Η γνωμοδότηση που υπέβαλα στην Επιτροπή είχε πολύ μεγάλο περιορισμό σε ό,τι αφορά τον αριθμό των χαρακτήρων, των γραμμάτων και την έκταση. Γι' αυτό έχει και τόσο συνοπτική μορφή. Πάντως θα συμπληρώσω αυτή τη γνωμοδότηση μέχρι τις 7 του μηνός, που είναι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και περιμένω και τα σχόλια των συναδέλφων. Πάντως ήδη είχαμε κάποια προκατακτική ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να προτείνουμε εναλλακτικού δείκτες και τις προτάσεις μας θα τις αποστείλουμε στην αρμόδια κατουσία επιτροπή που είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ που τα το λόγο, ο Λάμπερτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω τα σχόλιά μου με μία παρατήρηση. Παρατηρώ πόσο αραιό είναι το ακροατήριο σήμερα. Χθες ή προχθές συζητήσαμε στην Οικονομική ε, Επιτροπή τους περιβαλλοντικούς ε, λογαριασμούς, που είναι παρεφερές θέμα με το σημερινό. Και αντίστοιχη κατάσταση είχαμε ένα απόνα κροατήριο ουσιαστικά. Πολύ δυσάρεστη αυτή η κατάσταση, γιατί μπορεί αυτό το θέμα εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ανιαρό, αλλά είναι πολύ σημαντικό, γιατί το ΑΕΠ ουσιαστικά είναι αυτό που καθοδηγεί τις πολιτικές δεκαετίες ολόκληρες στην Ευρώπη. Και εφόσον αυξάνεται το ΑΕΠ, ε, αυξάνεται και η ευημερία. Αυτό είναι ένα αυτόματο συνειρμό. Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όταν το ΑΕΠ είναι υψηλό και το βιωτικό επίπεδο είναι υψηλό. Δυστυχώ τα τελευταία χρόνια και η πείρα μα έδειξε ότι ο σύνδεσμο μεταξύ τη αύξηση του ΑΕΠ και της ε, αύξηση των θέσεων εργασία ε, δεν είναι αυτόματο. Γιατί άλλο ΑΕΠ και άλλο ανάκαμψη ούτε αυξημένο επισημένη σημαίνει εξισορρόπηση των ανισοτήτων. Επίσης και ο, ο, ρόλος του ΑΕΠ σε ό,τι αφορά ε, τη κατανάλωση, εκεί υπάρχει σύνδεσμος. Υπάρχουν όμως προβλήματα και στις τρεις αυτές διαστάσεις. Σίγουρα η μετάβαση από το ΑΕΠ σε κάτι που θα περιλαμβάνει και άλλους δείκτες, θα είναι χρονοβόρα διαδικασία γιατί προϋποθέτει μια αλλαγή της πολιτικής κουλτούρας, ακόμη και της ε, υποσυνείδητης παιδείας του, του κόσμου, των πολιτών. Θα χρειαστεί χρόνος λοιπόν για να περάσουμε σε μια εποχή που θα λαμβάνει υπόψη και άλλα όργανα μέτρησης πέραν του ΑΕΠ, αλλά χρειάζεται να προσπαθήσουμε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τα σχόλιά τη και έχω να κάνω και εγώ ορισμένε παρατηρήσεις. Καταρχήν θα πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονό ότι αυτό το όργανο στόχο έχει να γίνει ένα, ε, να γίνει ένα όργανο για την λήψη, για τη χάραξη πολιτικών. Γιατί η μέτρηση της προόδου πέραν του ΑΕΠ δεν είναι αυτός σκοπός. Αυτός σκοπός είναι να σημειώσουμε πρόοδο και γνωρίζουμε ότι για την οικονομική διακυβέρνηση εξετάζουμε τα ελλείμματα, εξετάζουμε το χρέος και στην συζήτηση που είχαμε τη Δευτέρα με τον Όλυ Ρεν, είπε ότι σε αυτή τη φάση δεν θα είναι βέβαια δεσμευτικό, δεν θα είναι υποχρεωτικό, αλλά είναι ανοιχτό στην προσθήκη και άλλων δικτών κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Και σε αυτή τη γνωμοδότηση θα πρέπει να, δούμε, να πούμε ότι αυτοί οι νέοι δείκτες θα πρέπει να εξυπηρετήσουν την οικονομική διακυβέρνηση και να ενταχθούν στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης. Επίσης, γνωρίζουμε ότι ο τρόπο που καταμετράται σήμερα το ΑΕΠ δεν είναι ικανοποιητικό. Θα πρέπει να κρατήσουμε το ΑΕΠ ως όργανο ε, μέτρησης, αλλά να το καθαρίσουμε κάπως. Γιατί περιλαμβάνει και ε, καταστροφικά στοιχεία. Για παράδειγμα, με τις πετρελοκυλίδες ή με τους καρκίνους μπορεί να αυξάνεται το ΑΕΠ, αλλά θα πρέπει να το καθαρίσουμε από αυτά τα αρνητικά στοιχεία. Επίσης, Ξέρω ότι είμαστε Επιτροπή Βιομηχανίας κατά κανόνα, οπότε μας ενδιαφέρουν ε, ποσοτικά στοιχεία και όχι ε, γενική πολιτική θεώρηση. Αλλά θα πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη συγκέντρωσης δεδομένων. Δεδομένων που θα μας βοηθήσουν να βρούμε τους δείκτες και στο περιβαλλοντικό τομέα και στον κοινωνικό τομέα. Και απευθύνουμε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φροντίσει η Eurostat να αρχίσει να, μαζε... να συγκεντρώνει περισσότερα στοιχεία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δώσουμε κάποιους προσανατολισμούς ενδεκτικά για κοινωνικούς δείκτες για παράδειγμα. Ε, για θέμα το συντελεστής ε, ισότητας φύλων για παράδειγμα είναι σημαντικό για να δούμε τι ανισότητες υπάρχουν στην κοινωνία. Επίσης το θέμα της ένδυας ή της, ε, της υγείας. Δεν λέω ότι θα είναι εξαντλητικός αυτός ο κατάλογος των κοινωνικών δικτών, αλλά να αναφέρουμε αυτές τις προτάσεις ως ε, κατευθυντήριες γραμμές, ως προσανατολισμούς. Και για, το, για τις περιβαλλοντικές μετρήσεις γνωρίζουμε και από την πρωινή συζήτηση ότι η ενεργειακή απόδοση, απόδοση είναι πολύ σημαντική και η απόδοση των πόρων. Βέβαια δεν είναι εύκολο να καταμετρηθεί η ενεργειακή απόδοση ή η απόδοση πόρων μιας κοινωνίας. Αν όμως είμαστε σοβαροί και θέλουμε να έχει κάποιο ρόλο η Επιτροπή μας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε και τέτοια στοιχεία. Επίσης, υπάρχουν τα net adjusted savings ή το οικολογικό αποτύπωμα. Το οικολογικό αποτύπωμα δεν έχει ακόμη σωστό ορισμό. Χρειάζεται μια βελτίωση του ορισμού του οικολογικού αποτυπώματος. Αλλά ίσως αυτό είναι ένα σημείο αφετηρίας για να προβούμε και σε περιβαλλοντικούς δείκτες. Να συγκεκριμενοποιήσουμε λοιπόν κάπως τα πράγματα και να δώσουμε κάποιες συστάσεις εκ μέρους της Επιτροπής μας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος. γιατί επειδή είμαστε επιτροπή που ενδιαφέρεται για στοιχεία, θα πρέπει τέτοιου είδους ε, απτά σχόλια να υποβάλουμε προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα συντάξω και τροπολογίες σχετικές, γιατί δεν θέλω να αφήσουμε όλο το βάρος στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ, συνάδελφος το λόγο. Ευχαριστώ. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τι δύο τελευταίε εισηγήσεις, τη και θα ήθελα να θέσω το εξή ερώτημα. Αυτή η πολιτική ποιον εξυπηρετεί, αυτή η πολιτική την οποία θέλετε να ασκήσουμε, ποιον εξυπηρετεί. Πρωτίστως, τι οικολογικά προσανατολισμένε μη κυβερνητικέ οργανώσει, του consultants, ίσω τι νέε υπηρεσίε ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να, ιδρύσουμε αν θέλουμε να ερευνήσουμε αυτούς τους δείκτες μια τεράστια γραφειοκρατία εξυπηρετούν. αυτόν που δεν εξυπηρετούν είναι τις σοβαρές περιοχές της Ευρώπης και με την προσέγγιση αυτή απομακρύνεστε από την αρχή της ε, επικουρικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να σας εξηγήσω τι εννοώ. Δέχομαι την επιχειρηματολογία σας σε ό,τι αφορά την χωροταξία στα εθνικά κράτη-μέλη, σε ό,τι αφορά τις προστατευόμενες ε, φυσικές περιοχές, καταλαβαίνω τι λέτε για τους άξονες ανάπτυξης κτλ. Σύμφωνο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, και να συμπεριλάβουμε πιο έντονα περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς ε, τομείς. Αλλά αυτό που δεν αποδέχομαι είναι το εξή. Όταν μιλάμε για τον ορισμό περιοχών προώθησης, το ΑΕΠ ως τώρα αποτελεί μια αποδεκτή βάση μέτρησης ε, της αδυναμίας, αν θέλετε, ή μη μιας περιοχής. Και για να δούμε σε σοβαρά την σκέψη που εκφράζεται, αναφέρω κυριολεκτικά το σημείο 3 της γνωμοδότησής σας, κυρία εισηγητρία. Αναφέρει ότι για να επιτύχει η Ένωση του στόχου της την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ξενικονόμηση ενέργειας ε, προαπαιτεί μείωση του ΑΕΠ. Αυτό, μας τα σοβαρά, αυτός είναι ο πολιτικός σας στόχος. Θέλετε με τέτοιο τρόπο να στρεβλώσετε την ευρωπαϊκή πολιτική και να αφαιρέσετε από τις φτωχές περιοχές της Ένωσης ε, τέτοια υποστήριξη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πάρα πολύ επικίνδυνη αυτή η προσέγγιση που, μπορεί να, που προτείνεται, που δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό των ε, περιοχών αυτών. Η Ρινανία, το Ρουργκεμπίτ στη Γερμανία. Έχουμε μεγάλη εξόρυξη άνθρακα και με μεγάλα περιβαλλοντικά ε, περιβαλλοντική ζημιά. Με τα δικά σας κριτήρια θα παίρναμε κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία δεν χρειαζόμαστε. Και μια περιοχή η οποία είναι φτωχή στην Ανατολική Ευρώπη δεν θα έπαιρνε τα κονδύλια αυτά που τα παίρνει τώρα. Κυρίε και κύριοι, έχουμε και την στρατηγική το 2020, όπου αναφέρουμε ότι κάποια κονδύλια στα πλαίσια της στρατηγικής αυτής ε, αφιερώνονται ειδικά σε κάποιες φτωχές περιοχές σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά σας παρακαλώ μην στρεβλώσετε τις προσεγγίσεις αυτές της ε, αρχές της αλληλεγγύης που έχουν διαμορφωθεί μέσω από δεκαετίες ευρωπαϊκής πολιτικής. Ευχαριστώ να δώσω το τηλέφωνο στον συνάδελφο Κάμπος. Ε, ε, Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και πολύ χρήσιμο σε σχέση και με την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και όπως είπαμε, το θέμα αυτό έχει άμεση σχέση με την οικονομική διακυβέρνηση. Οπότε είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη συζήτηση και επίκαιρη. Θα ήθελα να συγχαρώ και την Επιτροπή για την ε, έκθεσή της, που είναι ένας τρόπος καταμέτρησης της πρόοδου πέραν της υλικής πτυχής μόνο της οικονομικής ανάπτυξης. Δεν θα πρέπει να ξεφύγουμε από τα κοινοτικά κείμενα, αρκεί να δούμε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020, για να διαπιστώσουμε πόσο ε, καινοτόμα είναι η Ευρώπη σε ό,τι αφορά την ε, υποβολή κάποιων προτάσεων για να αλλάξουμε τον κόσμο. Και θα πρέπει να, να προσαρμόσουμε στην καινοτομία και το οπλοστάσιο των δικτών μας. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε τους υπάρχοντες δείκτες με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς δείκτες, με πιο έγκυρη πληροφόρηση, με πιο ακριβείς δείκτες ό,τι αφορά την κατανομή των ανισοτήτων, να δημιουργήσουμε μηχανισμούς αξιολόγησης της βιώσιμης ανάπτυξης και να διευρύνουμε τους εθνικούς λογαριασμούς προκειμένου να περιλαμβάνουν και κοινωνικούς δείκτες, ε, θέματα απόδοσης ή περιβαλλοντικά. Ε, βέβαια, μερικές φορές έχουμε την αίσθηση ότι ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας, γιατί οι δείκτες για να είναι χρήσιμοι θα πρέπει να πληρούν μια σειρά προϋποθέσεων για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι έγκυροι πρώτα απ' όλα. Δηλαδή θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Επίσης θα πρέπει να είναι αξιόπιστοι. Θα πρέπει να είναι εύκολο να συλλεχθούν. Και θα πρέπει να είναι και σχετικά φθηνοί, να υπάρχει αντιστοιχεία σωστή κόστου ωφέλου. να είναι συγκρίσιμοι, να είναι επίκαιροι. και να είναι και εύρωστοι στη στεναρή. Γιατί η φιλοδοξία όλων που ασχολούμαστε με, ποσοτικά, με ποσοτικές μετρήσεις είναι ότι χρειαζόμαστε εύρωστους δείκτες. Σε όλους τους τομείς ε, το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού. Και έχω μία μικρή αφιβολία ως προς τη γνωμοδότηση της ε, αγαπητής Μαρίζα. Είναι ότι έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είπε ο συνάδελφος, ότι υπάρχει κίνδυνος ε, αύξηση της γραφειοκρατίας και κακής ποιότητας των δικτών, αν αρχίσουμε τώρα να ε, υποβάλουμε μια πληθώρα ε, δικτών που δεν χαρακτηρίζονται όμως από ακρίβεια, από ποιότητα ή δεν είναι εύρωστοι. Προσοχή λοιπόν να μην καταλήξουμε σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο δικτών. Θέλουμε ένα οπλοστάσιο δικτών, αλλά όχι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο ρητών. Επίσης, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα βασικά κενά. Και φάνηκε ότι το, στην στρατηγική του 2020 ότι το βασικό κενό είναι η ενημέρωση. Και θα πρέπει πρώτα απ' όλα να επικεντρώσουμε τους δείκτες που μας λείπουν σε θέματα απασχόλησης. Η απασχόληση θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης. Δεν είναι μια απλή συνέπεια η απασχόληση που βρίσκεται απλώς στο περιθώριο της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά θα πρέπει να βρεθεί στη καρδιά της οικονομικής ανάπτυξης. Και ευχαριστώ την εισηγήτρια για την ευκαιρία που μας έδωσε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριο Λάμπερτς και πάλι να απαντήσω στον συνάδελφο. Αλλά ξέχασα το όνομά σα. Πολύ λυπάμαι. Να πω δύο λόγια. Καταρχά, όταν λέτε ότι αν σταματήσουμε να μετράμε άλλα στοιχεία, αυτό σημαίνει περαιτέρω γραφειοκρατία, πρέπει να σα πω ότι δεν σύμφωνο. Μετά αποδέχομαι αυτό σε επιχείρημα. Φυσικά υπάρχει ο κίνδυνο αυτό, αλλά θα πρέπει να το αποφύγουμε αυτό. Και γι' αυτό αναφέρθηκα ειδικά στη Eurostat. Έχουμε μια υπηρεσία η οποία συλλαγεί ε, στατιστικά στοιχεία, η οποία έχει αποδειχτεί και αποτελεσματική όπου της έχει επιτραπεί να δρά. Φυσικά, αν κάποιες χώρες κλείνουν την πόρτα, αυτό δυσκολεύει το έργο της, αλλά υπάρχει μια υπηρεσία η οποία είναι υπεύθυνη για τέτοια συλλογή στοιχείων. Δεν ε, συνηγορώ υπέρ της δημιουργίας άλλης υπηρεσίας. Κατά δεύτερον, αμφισβητείται κατά πόσο υπάρχει ανάγκη να μετρούνται και άλλα στοιχεία να κάνω μια σύγκριση με το αυτοκίνητό σας. Όταν οδηγείτε, θέλετε να ξέρετε πόσο καύσιμο έχει ακόμα στο αυτοκίνητό σας. Αν δεν το μετράτε αυτό, θα βρεθείτε προεκπλήξεως, δυσάρεστης. Γιατί λοιπόν το εξετάζουμε αυτό, γιατί θέλουμε να ξέρουμε αν οι πόροι που χρησιμοποιούμε εξαντλούνται. Για παράδειγμα, να σας πω ότι και ο πατέρας μου δεν ε, μπορούσε να μετράει με το αυτοκίνητό του πόσα ε, χιλιόμετρα είχε κάνει. Εγώ έχω τέτοιο μετρητή στο αυτοκίνητό μου και έτσι μπορώ να μετρήσω πόσο καύσιμο ξοδεύω και να προσαρμόσω την οδηγική μου συμπεριφορά. Αυτό το ίδιο λέμε. Δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμη αυτή η δυνατότητα χρειάζονται περισσότερα στοιχεία πέρα από την ταχύτητα, για παράδειγμα, στο αυτοκίνητο, στο αεροπλάνο και το καθεξής. Είπατε ότι αυτό θα έχει αρνητική επίπτωση στην, ε, στην αλληλεγγύη λόγω των ε, ταμείων, των διορθωτικών σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να κινηθούμε προ την κατεύθυνση αυτή. Είμαστε υπέρ τη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και φυσικά αποτελούν εργαλείο σημαντικό προς την κατεύθυνση αυτή τα διευθυντικά ταμεία. Αν έτσι λοιπόν κατανοήσατε τις προτάσεις μας, ίσως δεν εκφράστηκα καλά. Αλλά ειλικρινά δεν αποτελεί αυτό πρόταση των πράσινων. Δεν θέλουμε τίποτα ρεξικέλευτο να προσθεθούν κάποιοι δείκτες όπως για παράδειγμα για το 2020 αναφέρεται στοιχεία για τη φτώχεια. Ανέφερα για παράδειγμα την χρήση των πόρων. Προφανώς λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε προς μια τέτοια κατεύθυνση. Ευχαριστώ και το λόγο έχει και πάλι η η κυρία Ματίας. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Ήδη από τα σχόλια φάνηκε πόσο σημαντική είναι η σημερινή συζήτηση από πολιτική άποψη για το πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε τη μέτρηση της πρόοδου με δείκτες πέραν του ΕΠ. Όπως είπα και στην αρχική μου παρουσίαση, Επειδή περιοριζόμουν στο ότι φορά την έκταση και το έβρισκο γνωμοδότηση, δεν μπόρεσα να επεκταθώ και να είμαι πολύ πιο συγκεκριμένη, γιατί οφείλουμε να τηρούμε τις διατάξεις. Γι' αυτό και θα, όπως σας είπα, θα υποβάλω τροπολογίες για να καταθέσω και πιο απτές προτάσεις για τους δείκτες. Έχω και κάποια άλλα σχόλια σχετικά με τη συζήτηση που έγινε. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι το ΑΕΠ ως όργανο μέτρησης είναι ανεπαρκές. Αυτή η συζήτηση δεν είναι καινούρια. Ξεκίνησε πριν από χρόνια. Και η πρόταση της Επιτροπής, ε, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πιστεύω ότι είναι επίκαιρη, είναι πολύ σωστή και πολύ εύστοχη και έχει σημαντικές προτάσεις. Γι' αυτό και καλό θα ήταν και εμείς να τις συμπληρώσουμε και να τους δώσουμε μια πιο συγκεκριμένη προοπτική. Πάντως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι ένα ακόμη βήμα σε μία σειρά προσπαθειών που έγιναν για να θεσπιστούν συμπληρωματικοί δείκτες που θα καταμετρούν καλύτερα το βιωτικό επίπεδο και την ευημερία των πολιτών και θα αντικατοπτρίζουν καλύτερα την πραγματικότητα της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Μία σειρά θεσμών και Ινστιτούτων προσπάθησαν ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ΟΗΕ, να θεσπίσουν τέτοιους συμπληρωματικούς δείκτες και έγιναν και συνδιασκέψεις ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να γίνει η ανάλυση αυτού του θέματος. Όταν περνάμε λοιπόν τόσα χρόνια και προτείνονται τόσοι διαφορετικοί συμπληρωματικοί δείκτες για να καταμετρηθεί η ποιότητα της ζωής και οι κοινωνικές ε, συνθήκες για να υποστηριχθούν καλύτερα και να ληφθούν πιο τεκμηριωμένες οικονομικές ε, αποφάσεις. Αφού γίνονται τότε λοιπόν συζητήσει, σημαίνει ότι τα υπάρχοντα όργανα μέτρησης και κυρίως το ΕΠ δεν αρκούν. Γι' αυτό θα προτείνουμε εναλλακτικά μέτρα. Είναι σαφής η ανάγκη αυτή και θέλουμε να υποβάλουμε συμπληρωματικούς δείκτες που θα κάνουν την μέτρηση πιο αξιόπιστη και πιο ακριβή. Δεν είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε εδώ ένα γραφειοκρατικό τερατούργημα και να περιπλέξουμε τη ζωή μας. Δεν ήταν ε, σε καμία περίπτωση αυτή η πρόθεσή μου να επιτείνω την γραφειοκρατία ή να αλλοιώσω την αξιοπιστία ενός οργάνου μέτρησης. Ίσα ίσα εγώ θεωρώ ότι χρειαζόμαστε τους δείκτες και όργανα μέτρησης, αλλά ακριβώ αυτή την αδυναμία έχει το ΑΕΠ ότι δεν είναι αρκετά αξιόπιστο και αντιπροσωπευτικό όργανο μέτρησης. Μην ξεχνάτε ότι διανύουμε μια βαθύτατη οικονομική και κοινωνική κρίση σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Οπότε Έχω την αίσθηση ότι για να καταμετρήσουμε την επιτυχία των οικονομικών πολιτικών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πέραν του ΑΕΠ την πραγματική κοινωνική πραγματικότητα και τις πραγματικές κοινωνικές ανισότητες. Τέτοιου είδου κριτήρια θα πρέπει να, θα χρησιμοποιήσουμε για να αποτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα των οικονομικών πολιτικών και όχι μόνο το ΑΕΠ. Φυσικά θα κληθούμε να κάνουμε και κάποιες επιλογές. Αναφέρθηκε ότι η στρατηγική του 2020 δίνει κάποιες κατευθύνσεις για τους λογαριασμούς, για τη διεύρυνση των εθνικών λογαριασμών. Το θέμα των κοινωνικών κριτηρίων και των περιβαλλοντικών είναι επίσης ε, πολύ σημαντικό. Είναι θεμελιώδους σημασίας. Αλλά δεν πρόκειται να ανοίξουμε κανένα κουτί της Πανδώρας, ούτε πρόκειται να δημιουργήσουμε ένα γραφειοκρατικό τέρας. Ήδη υπάρχουν ε, συστήματα συλλογή συγκέντρωση πληροφοριών. Απλώς θα συμπληρώσουμε το ΑΕΠ με άλλους δείκτες, ώστε να καταλήξουμε σε πολύ πιο αξιόπιστους τρόπους μέτρησης γιατί το ΑΕΠος μοναδικό όργανο δεν αρκεί. Και θα πρέπει φυσικά να κάνουμε και κάποιες επιλογές. Υπάρχουν κάποιοι πολυδιάστατοι δείκτες και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε. Οι επιλογές μας θα πρέπει να γίνουν μέσω του δύσκολου εγχειρήματο των διαστάσεων που θα επιλέξουμε. Και θα πρέπει να δούμε τι θα βάλουμε στην καρδιά του όλου εγχειρήματος πέραν του πλούτου και πέραν του ΑΕΠ, ποιον άλλο δείκτη θα βάλουμε στο επίκεντρο του προβληματισμού. Τα περιβαλλοντικά θέματα, τα κοινωνικά θέματα, την απασχόληση. Και αυτοί οι παράγοντες θα πρέπει να βρεθούν στο κέντρο της αξιολόγησης. Πιστεύω ότι η συζήτηση γίνεται για να ενισχύσουμε την ακρίβεια των μετρήσεών μας και να κάνουμε πιο εύρωστη την αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής. Η συζήτηση αυτή γίνεται για να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τη μέχρι τώρα κατάσταση. Γιατί έχουμε ένα μέτρο μακροοικονομικής δραστηριότητας που αγνοεί τους μη εμπορικού παράγοντες. Δεν μπορούμε να αποκλείουμε τελείως τους μη εμπορικού παράγοντες. Γιατί έτσι καταλήγουμε σε συμπεράσματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ούτε από κοινωνική, ούτε από περιβαλλοντική άποψη και ούτε από άποψη απασχόλησης. Äh, Σα ευχαριστώ. Δεν τα κανεί άλλο το λόγο. 7 Οκτωβρίου λοιπόν είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών και περνάμε στο 17α. Θα συζητούσαμε το κείμενο το οποίο σας έχουμε ήδη αποστείλει. Δεν ξέρω βέβαια αν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Θέλετε το λόγο να το σχολιάσετε. Συνάδελφε, δεν χρειάζεται. Την επιστολή, την επιστολή που απεστήλαμε ως ομάδα στην ε, Επιτροπή περιβάλλοντος. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτά που συμφωνήσαμε έγραψα. Αν δεν θέλει κανείς να πάρει το λόγο, να προχωρήσουμε. Ναι, ναι, άμα δεν ε, μιλήσει κανείς θα προχωρήσω. Στο 18 της ημερήσιας διαταξής παρουσίαση της μελέτης με θέμα αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας. Να καλωσορίσω τους ομιλητές μας. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Okay. Η κυρία Καβάλιο θέλει να πάρει το λόγο στην επιστολή, για την επιστολή. Έχετε το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το θέμα του Κανκούν. Λυπούμε που το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος δεν επέτρεψε επισήμως και την ανάμεξη της Επιτροπής Ήτρε και ελπίζω την επόμενη φορά να εμπλακούμε σε προγενέστερο στάδιο γιατί το θέμα των κλιματικών αλλαγών αφορά και την βιομηχανία, την Επιτροπή Βιομηχανίας ενέργειας. Και καλό θα ήταν να εμπλεκόμαστε στον ίδιο βαθμό με την Επιτροπή Περιβάλλοντος για τα θέματα κλιματικών αλλαγών που μας ενδιαφέρουν εξίσου. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που υποστηρίζουν και οι υπόλοιπε ομάδες. Οι ομάδες αποφάσισαν να συνυπογράψουν ένα συμβαστικό κείμενο και θα είναι πολύ σημαντικό οι ομάδες να συμπαρασταθούν ε, και να, συν, να συμφωνήσουν ως προς το κείμενο που θα πρέπει να στείλουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα πρέπει να είναι ενιαίο αυτό το κείμενο για να είναι πιο στεναρή η θέση που θα δώσουμε ως Επιτροπή Ήτρε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ζητούμε βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, ζητούμε μια διεθνή συμφωνία που θα εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και συνθήκες θεμητού και ίσου ανταγωνισμού στις εντατικές άποψη άνθρακα βιομηχανίες. Επίσης, αναφέραμε και την προσθέμενη αξία της εξοικονόμησης ενέργειας στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Αυτή θα είναι πολύ σημαντική συμβολή για την υλοποίηση των στόχων μείωσης του διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ κυρία Καρβάλιο να επαναλάβω ότι δεν ήταν δίκαιο ο τρόπο που μας αντιμετώπισε η Επιτροπή Περιβάλλοντος ω τώρα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούμε να τον εξαναγκάσουμε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με την έκθεση για το πετρέλαιο είναι η διάσκεψη των Προέδρων να παρέμβει. Ως τώρα δεν έχει ταχθεί υπέρ μας η διάσκεψη των Προέδρων και εξαρτάται από εμάς το τι θα κάνουμε σε ό,τι αφορά την έκθεση για το πετρέλαιο. συμφωνήσαμε να συμμετάσχει η Ήτρε και για το COP16 παρόμοια, παρόμοια ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ουσιαστικά είναι ε, αλληλοσεβασμού. Και να περάσουμε λοιπόν στο 18. Θα έχετε μπροστά σας τα έγγραφα, τη μελέτη που την έχουμε στη διάθεσή μας εδώ και κάποιο καιρό. Ο Ζαν Κριστόν Πλανουά και ο Ντέιβιτ Έλισον είναι μαζί μας σήμερα και θα μας παρουσιάσουν εν συντομία τα πορίσματα της μελέτης. Είχατε και έχετε μπροστά σας τα έγγραφα αυτά. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να προσέξετε την παρουσίαση αυτή και να θέσετε ερωτήματα. Όσοι έχετε απομείνει στην αίθουσα τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ και σας δίνω το λόγο. Δεν ξέρω ποιο από τους δύο θα ξεκινήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω. Ευχαριστώ που μας ε, προσκαλέσετε εδώ σήμερα και που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τα πορίσματα της μελέτης αυτής. Σαν Κριστόφ Λανουά ονομάζομαι. Δουλεύω για μια ε, εταιρεία βιώσιμης ενέργειας και βλέπετε ποιοι είναι αυτοί που συνέβαλαν στην μελέτη για την αποκέντρωση της παραγωγής της ενέργειας. Την ξεκίνησε ο Ματίας Χάρτμαν από τη TLSP και από το Κολέγιο της Ευρώπης, από τον David Ellison, τον συναδελφό μου. Συμμετείχε και αυτός, το VTT, Τεχνικό Κέντρο της Φιλανδίας, έρευνας και η όλη εργασία αναθεωρήθηκε από τον Πέτρο Λινάρες από το Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης. Σκοπός της ε, μελέτης είναι να, ήταν να εκτιμηθεί η οικονομική και τεχνική κατάσταση της ε, αποκέντρωσης της παραγωγής ενέργειας στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει. Προτείναμε λοιπόν ε, κάποιες πολιτικές συστάσεις σε ό,τι αφορά α, τις επενδύσεις, την τεχνολογική ανάπτυξη, τις επενδύσεις, τα συγκεκριμένα μέτρα για τις ε, ε, μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις και τον τονισμό των προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η βασική ιδέα πίσω από την μελέτη αυτή ήταν η εξής. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μία φάση πρωτοφανών αλλαγών σε ό,τι αφορά την διοργάνωση των συστημάτων της. Ε, κινούμαστε από τα αριτά καύσιμα και από το σύστημα πυρηνικών καυσίμων σε ένα σύστημα πιο αποκεντρωμένο σε ό,τι αφορά την παραγωγή ενέργειας. Εξαρτώμαστε όλο και πιο πολύ από ανανεώσιμες πηγές και το σύστημα πιο πολύ από ανταπόκριση στις υφιστάμενες ανάγκες. Όλα αυτά θα τα κοιτάξουμε και αργότερα. Όλα αυτά λοιπόν ε, προέρχονται από κάποιες ενιστώσεις τις οποίες αναφέρω εδώ σε διαφάνεια. Καταρχάς, ό, όταν ε, εγκρίνατε τους στόχους για το 2020, αυτό το υπερλαμβάνει μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, αύξηση του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζουμε την ε, ασφάλεια εφοδιασμού και η ανανεώσιμη οι ανανεώσιμες ενέργειας μπορεί κάποιες στιγμές να περιορίζουν την Ένωση και την παραγωγή ενέργειας και θα πρέπει να φροντίσουμε να αποτραπούν ενδεχόμενα blackout για παράδειγμα. Από την άλλη, η ζήτηση για ρεύμα αυξάνεται και στο τρίτο πακέτο για την ενέργεια βλέπουμε ότι απελευθερώνονται οι ενεργειακές αγορές. Ας περάσουμε τώρα σε κάποιους ορισμούς. Καταρχάς, καταναμημένη παραγωγή. Πρόκειται για τις ε, μικρής κλίμακας ικανότητες που συνδέονται στο δίκτυο διανομής κατευθείαν χαμηλού και μεσαίου βολτάζ. Η πρώτη βασική πηγή ενέργειας είναι σε πολλές περιπτώσεις ανανεώσιμες και διατίθεται σε τοπικό επίπεδο. Μιλάμε λοιπόν για φωτοβολταϊκά, θερμικά, αιωλικά για CHP, συνδυασμένη δηλαδή θερμική και, ολική, και ηλιακή ενέργεια και ωκεανική ενέργεια, είτε από βιομάζα, είτε από ρηκτά καύσιμα, από φυσικό αέριο. Δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι το demand response, η ανταπόκριση στη ζήτηση. Μιλάμε για την έξυπνη διαχείριση της ενεργειακής χρήσης από πλευράς καταναλωτή. Δεν ε, μιλάμε απαραίτητα για εξοικονόμηση ενέργειας, μάλλον για την μετατόπιση του φορτίου ενέργειας χρονικά. Να διασφαλίσουμε δηλαδή, για παράδειγμα, ότι δεν ξεκινάει το πλυντήριο στις 6 το απόγευμα, που είναι ε, ώρα υψηλή ζήτηση ρεύματο, αλλά ίσως δύο-τρει ώρε μετά, όταν θα έχει περιοριστεί κάπω η Και Ως απάντηση σε αυτές τις πρωτοφανείς αλλαγές, το δίκτυο, το ηλεκτρικό, θα πρέπει επίσης να προσαρμοστεί, να αλλάξει, να κινηθεί προς μια πιο ενεργή, αν θέλετε, μορφή. Smart Grid, έξυπνα δίκτυα, έτσι τα ονομάζουμε. Τα έξυπνα δίκτυα δεν έχουν ακόμα πλήρως και ρητά οριστεί τι σημαίνει όμως, τι σημαίνουν αποκέντρωση της ε, παραγωγής ενέργειας, έξυπνη διαχείριση της ενέργειας και της ε, ενεργειακής αποδοτικότητας. Μία άλλη σημαντική έννοια είναι η αποθήκευση ενέργειας. Οι ανανεώσιμες ε, ενέργειες δεν είναι σταθερές ως προς την παροχή Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα λοιπόν αποθήκευσής τους για να τις χρησιμοποιεί κανείς όταν τις χρειάζεται. Θα υπάρχει λοιπόν όλο και μεγαλύτερη ανάγκη αποθήκευσης ε, των ε, ενεργειακών αυτών μορφών. Κάτι τελευταίο πολύ σημαντικό είναι ο ρόλος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα αποκεντρωμένα συστήματα ενέργειας εκπροσωπούν περίπου το 30% της ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρώπης. Και είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης σε ό,τι αφορά την ε, κατανάλωση και τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να συμπεριληφθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε οποιοδήποτε πολιτική σε οποιοδήποτε πλαίσιο πολιτικής που αφορά την ενεργειακή κατανάλωση. Να σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία εντάχει η υδροελεκτρική ενέργεια αποτελεί με μεγάλη διαφορά τη μεγαλύτερη μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αιωλική ενέργεια είναι η δεύτερη και η Ευρώπη είναι κορυφαία σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις ε, αιωλικής ενέργειας. Μας, έχει όμως ξεπεράσει, μας έχουν ξεπεράσει η ΕΠΑ και η Κίνα το CHP επίσης ε, ανταποκρίνεται σε μεγάλο ποσοστό της ηλεκτρικής ε, κατανάλωσης και άλλες τεχνολογίες όπως τα φωτοβολταϊκά, τα ηλιακά θερμικά και η ωκεανική ενέργεια είναι ε, πολύ μικρής, πολύ μικρής συμμετοχής. Και τις επόμενες διαφάνειες θα σας παρουσιάσει ο Ντέιβιτ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια για το γιατί μας απασχολεί η αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας. Καταρχάς, επειδή μπορεί να αποτελέσει βασικά στοιχεία για τα μελλοντικά δίκτυα, γιατί ένα από τα προβλήματα που έχουμε με τις τρέχουσες ε, ε, ανανεώσιμες ενέργειες οι οποίες δεν είναι μόνιμες είναι ότι δημιουργούνται μποτιλιαρίσματα σε ό,τι αφορά την ε, παροχή ενέργειας. Ακριβώς επειδή δεν είναι μόνιμες οι πηγές αυτές. Υπάρχουν κάποιες ε, απαντήσεις, ε, για παράδειγμα το DR. Μια άλλη λύση είναι η καλύτερη διασύνδεση των χωρών, γιατί έτσι μπορεί να μεταφέρεται η ενέργεια μεταξύ μεγαλύτερων περιοχών. Και έτσι μπορεί να χρησιμοποιείται με μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Και φυσικά για να τα πετύχουμε όλα αυτά χρειάζεται πιο πολύ έρευνα, ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση στην ζήτηση και τις τεχνολογίες εφιών δικτύων, αλλά και για άλλες τεχνολογίες που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τι προαπαιτείται λοιπόν για τα αποκεντρωμένα συστήματα ενέργειας. Καταρχάς χρειάζεται μια ενσωμάτωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των δικτύων. Βασιζόμαστε λοιπόν σε αυτή την ιδέα της διασύνδεσης. Επίσης, ε, να πούμε ότι αν δεν είναι πλήρως ενσωματωμένα τα δίκτυα αυτά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερες δυσκολίες σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της ε, χρήσης ενέργειας. Όσο πιο πολύ ενσωμάτωση και ενοποίηση, τόσο το καλύτερο δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, σημαντικό είναι να υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο Αυτό θεωρητικά ρυθμίζεται από το τρίτο πακέτο ενέργειας. Και ένα βασικό ζήτημα είναι τα θέματα προτεραιότητας για τις ανανεώσιμες ενέργειες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση. Θα επανέλθω σε αυτό. Τρίτο στοιχείο χρειάζεται πιο συνεκτική και ευέλικτη νομοθεσία, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι αρκετή η ευελιξία που έχει να επιδείξει το πλαίσιο το νομοθετικό και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την πιο ευέλικτη αξιοποίηση των πόρων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι ανανεώσιμε. Τέλος, χρειάζεται μια διαφανής δομή σε ό,τι αφορά τα κίνητρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θα ήταν καλή ιδέα αυτό. Γιατί στην παρούσα φάση οι πιο πολλέ στρατηγικές για την πρόωθηση των επενδύσεων σε ό,τι αφορά τι ανανεώσιμε ενέργειε, βρίσκονται στα χέρια των κρατών μελών. Δεν υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Θα πρέπει να γίνουν πιο βραστήρια βήματα, αν θέλετε, προς την κατεύθυνση αυτή και πολλά μπορούμε να κάνουμε για να δοθούν τέτοια κίνητρα πανευρωπαϊκά. Τέλος, ένα βελτιωμένο δίκτυο πλαίσιο για την ε, έρευνα. Και αυτό θα απέβαινε προς όφελος της αποκέντρωσης της ενέργειας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση των δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο η για τα ανταπόκριση στις ανάγκες καθορίζεται βασικά από το μέγεθος του δικτύου. Όσο πιο μεγάλο είναι το δίκτυο, τόσο πιο εύκολο είναι να ρυθμίζονται να ρυθμίζεται η παροχή. Άρα, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο θα διευκολύνει μια πιο ενσωματωμένη, μια πιο ενεπιμενή διαχείριση της ενέργειας και αυτό φυσικά θα ε, έχει μεγάλο αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την ισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Θα πιο γρήγορη πρόοδο σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση μεταξύ των ευρωπαϊκών δικτύων, γιατί γίνεται με πρόοδος, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και μεγάλη υποστήριξη από το κοινό και χρειάζεται επίσης ε, στενή παρακολούθηση, γιατί πολλοί στόχοι έχουν ε, δηλωθεί, αλλά στην πράξη δεν επιτυχάνονται συνήθως. Θα μπορούσαμε με στενότερη παρακολούθηση να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της ε, πολιτικής. Αν δεν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο, δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπότε χρειάζεται ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που θα είναι και ευφυέ φυσικά δίκτυο, για να ξέρουμε πώς, τι ποσότητα ενέργειας ε, περνάει από το δίκτυο. Δεν είναι ευφυέ στο δίκτυο, δεν μπορούμε να μετρήσουμε την ποσότητα αυτή. Επίσης, πρόσβαση σε ένα τέτοιο πανευρωπαϊκό δίκτυο. Το τρίτο ενεργειακό πακέτο θεωρητικά ασχολήθηκε με το θέμα αυτό, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να εφαρμόσουν πολιτικές πρόσβασεις, δικές τους πολιτικές πρόσβασεις στο δίκτυο. Και φυσικά θα μπορούσαν να υπάρξουν σημαντικές διαφοροποιήσεις για το πώς γίνεται η διαχείριση της πρόσβασης στο δίκτυο από χώρα σε χώρα. Το βασικό θέμα είναι ποιος θα πληρώσει για τη διασύνδεση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο. Αυτός που θα παράγει την ανανεώσιμη ενέργεια με μια ανεμογεννήτρια ή το ίδιο το σύστημα του δικτύου ή οι διαχειριστές του δικτύου θα πληρώνουν αυτή τη διασύνδεση. Και πάλι υπάρχει μεγάλη διαφορά σε ό,τι αφορά το εύρος των επιλογών από χώρα σε χώρα. Αν θέλει κανείς πραγματικά να ενθαρρύνει τις ανανεώσιμες ενέργειες, τότε λογικό είναι να απαιτεί από τον διαχειριστή του δικτύου να πληρώσει τη διασύνδεση. Αυτό θα ήταν είδο ε, επιμερισμού, κοινωνικού επιμερισμού των δαπανών. Γιατί ένα τμήμα των αυξανόμενων δαπανών του δικτύου θα μετακυλιστεί στην τιμή της ενέργειας. Οπότε αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις ανανεώσιμες ενέργειες, ένας τρόπος είναι να μεταφέρουμε τη χρηματοδότηση για την πρόσβαση στο δίκτυο προς τον διαχειριστή του δικτύου, προς τον κύριο του δικτύου. Επίσης, ε, η εφαρμογή από τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιβλέπεται πιο στενά για να δούμε τι εύρος έχει αυτή η διαφοροποίηση και τι προσκόμματα υπάρχουν σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις ανανεώσιμες ενέργειες και τι στρατηγικές χρησιμοποιούν ή επιλέγουν τα διάφορα κράτη-μέλη. Επίσης θα μπορούσαμε να ε, ενισχύσουμε τις διατάξεις για την πρόσβαση στο δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερα αν υπάρχουν προβλήματα στην εφαρμογή σε συγκεκριμένες χώρες αλλά αυτό είναι θέμα που θα το εξετάσουμε αργότερα. Επίσης, ε, χρειαζόμαστε πιο ελαστικό νομοθετικό πλαίσιο και πιο συνεκτικό. Υπάρχει ένα πρόβλημα συμβατότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ε, ενεργειακή απόδοση και την οδηγία για το συνδυασμό θερμότητας και ηλεκτρισμού. πώς, με βάση την οδηγία CHP, τι ποσοστό ενέργειας θα παράγει, τι ποσοστό θερμότητας, ενώ η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων μιλάει για καλύτερη θερμομόνωση στα κτίρια. Οπότε Ίσως είναι αντιφατικές οι δύο γιατί η μία προβλέπει μεγάλη παραγωγή θερμότητας, ενώ η άλλη λόγω της θερμομόνωσης ίσως δεν ε, μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι ότι δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ελαστικότητα στο σύστημα εμπορίας εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους τομείς που δεν εμπίπτουν ε, στο σύστημα εμπορίας εκπομπών αποτελέσματα αυτής της αναλαστικότητας είναι ότι δεν υπάρχουν και πολλά ενάυσματα για να προωθηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτίριων. Δεν είναι δεσμευτική η στόχη για την ενεργειακή αποδοτικότητα, με εξαίρεση την οδηγία ESD που απαιτεί 9%. Και οι πρωτοβουλίες για την ενεργειακή απόδοση δεν συνδέονται με το ETS, την εμπορία εκπομπών, ή το ενεργειακό και περιβαλλοντικό πακέτο, το κλιματικό πακέτο. Μπορεί να δίνονται κάποια ενάψματα για την ενεργειακή απόδοση, αν η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια ε, οδηγήσει σε μόρια που μπορεί κανείς να αγοράσει, να πουλήσει στην αγορά εμπορίας, στην αγορά του συστήματο εμπορία εκπομπών, για παράδειγμα. Να υπάρχει μια τέτοια διασύνδεση. Αυτό θα ήταν ένα κίνητρο. Θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε αυτή, αυτού του είδους την ελαστικότητα, αλλά χωρίς τέτοια ελαστικότητα δεν είναι σαφές ότι θα γίνουν επενδύσεις ε, στους πιο αποτελεσματικούς κλάδους από άποψη κόστους-οφέλους. Οπότε μια αυξανόμενη ελαστικότητα θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να αυξήσει και τα κίνητρα για επενδύσεις σε περισσότερη ενεργειακή απόδοση και άρα και σε μείωση των εκπομπών. Σε ό,τι αφορά τα, τους μηχανισμούς των κρατών μελών για την πρόθεση των ανανεώσιμων ενεργειών, δύο κυρίως είναι τα ισχύοντα συστήματα στις χώρες μέλη. Υπάρχει το FIT, όπου ο παραγωγός της ανανεώσιμης ενέργειας πληρώνει ένα δασμό και υπάρχει και το σύστημα πιστοποιητικών, το RO, Renewable Obligation, που απαιτείται από τις εταιρείες που παράγουν ενέργεια να ένα τμήμα της ενέργειας που παράγουν να το παράγουν από ανανεώσιμες πηγές. Το πρόβλημα με τη στρατηγική για την υποχρέωση ανανεώσιμης ενέργειας έγκυται στο ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματική αυτή η στρατηγική όσο το σύστημα FIT, γιατί, του, του δασμού δηλαδή. Άλλωστε το σύστημα για την καταβολή δασμού ήταν πολύ πιο παλιό. Ένα άλλο από τα προβλήματα της ε, υποχρέωση ανανεώσιμη πηγή ενέργειας είναι ότι είναι πιο δαπανηρό. Ευνοεί τους ε, μεγάλους παραγωγούς, εις βάρος των μικρομεσαίων. Γιατί και στους μικρομεσαίους είναι πολύ δύσκολο, γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία ε, να μπορέσουν να συμμετέχουν στους πληροδοτικούς κανονισμούς. Επίση υπάρχουν διακοιμάνσει και στι ε, τιμέ τη ενέργεια. Γι' αυτό και δεν μπορεί κανεί να κάνει μακροπρόθεσμε προβλέψει του κέρδου των ωφελών. Οπότε αυτό είναι αντικίνητρο για συμμετοχή στο σύστημα. Και από τις, περιστάσεις, περιπτώσεις που είχαμε δεν, ε, δεν είχαμε πολύ καλά παραδείγματα. Μάλιστα χαρακτηριστικό παράδειγμα μικρής επιτυχίας ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το Ηνωμένο Βασίλειο που χρησιμοποιεί το σύστημα FIT. Πάντως υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών ανάλογα με το σύστημα που, το, χρησιμοποιούν. Το μπλε χρώμα είναι το σύστημα FIT, το κόκκινο είναι της υποχρέωσης ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και άλλες χώρες έχουν ένα μείγμα. Η Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, έχει σύστημα μεικτό, FIT και RO. γιατί το αρχικό σύστημα της ανανεώσιμης υποχρέωσης, υποχρέωσης ανανεώσιμης ενέργειας δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό και προσθέθηκε και μια πτυχή FIT. Σε ό,τι αφορά τα συστήματα FIT, γενικώ ήταν πιο επιτυχημένα και αρχίζουν και μετατρέπονται στον κανόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε ότι οι περισσότερες χώρες είναι χρωματισμένες με μπλε χρώμα, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούν ε, σύστημα FIT. Μπορούμε πια να προσθέσουμε και τη Φιλανδία σε αυτό το χρώμα γιατί μόλις ε, εγγενίασε για την πράσινη ενέργεια το σύστημα FIT. Χώρες που έχουν πιο μακρόχρονη πείρα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η Γερμανία, χρησιμοποιούν ε, παραδοσιακά το σύστημα FIT και μάλιστα η Γερμανία από τις χώρες που χρησιμοποιεί πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μάλιστα πολλοί λένε ότι αυτό έγινε χάρη στο σύστημα FIT αλλά και άλλες χώρες με νεότερα σημείωσαν επιτυχία, όπως η Ισπανία. Το πλεονέκτημα του συστήματος FIT είναι ότι ευνοούν την άμεση ένταξη των ανανεώσιμων ενεργειών. Επίσης ε, εξυπηρετούν και τους μικρούς, ε, ε, μεγάλους αλλά και τους μικρούς παραγωγούς. Μπορεί κανείς ακόμη και στο σπίτι του να εγκαταστήσει έναν ηλιακό θερμό και να, έχει, να παράγει μόνο στην ενέργειά του. Οπότε το σύστημα FIT είναι ευνοϊκό όχι μόνο για τους μεγάλους παραγωγούς αλλά και τους μικρούς. Και γενικώ στο σύστημα FIT υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια, βεβαιότητα και χαμηλότερο κόστος Βέβαια και πάλι υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών μελών και μάλιστα στην έκθεσή μας υπάρχουν πολύ πιο διεξοδικά στοιχεία. Αλλά είναι πολύ κοινό, ή τουλάχιστον γίνεται όλο και πιο κοινό, οι, οι τιμές να τη χάνουν εγγύηση για πολύ περισσότερα χρόνια, για μια εικοσαετία για παράδειγμα. Και αυτό είναι σημαντικό, να υπάρχει μια βεβαιότητα, γιατί κανείς όποιο χρησιμοποιεί το FIT βλέπει ότι για 20 χρόνια έχει εγγυημένη τιμή ενέργεια. Αυτό είναι πολύ ελκυστικό. Και γενικώ το κόστος ε, είναι χαμηλό. Δεν χρειάζεται κανείς να υποβάλει ε, αίτηση, ούτε να συμμετέχει σε διαγωνισμούς. Απλώς εγκαθιστά το σύστημα και πληρώνει την ενέργεια. Είναι πολύ πιο εύκολη η διαδικασία. Μία άλλη καλή ιδέα θα ήταν να έχουμε μία διαφανή πανευρωπαϊκή δομή κινήτρων. Καλό θα ήταν να έχει πανευρωπαϊκό χαρακτήρα αυτή η δομή. Γιατί δεν υπάρχει ισότητα σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες των χωρών και τα αποτελέσματα. Μερικές χώρες ήταν πιο επιτυχημένες, άλλες λιγότερο. Οπότε με ένα πανευρωπαϊκό σύστημα στρατηγικής και κινήτρων θα είχαμε μια μεγαλύτερη ομοιομορφία. Επίσης μπορούμε να υποστηρίξουμε και στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Γιατί τέτοιου είδους συστήματα αποθήκευσης χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις, ανάπτυξη, άρα και περισσότερα ενάψματα. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για αποθήκευση ενέργειας. Το θέμα του φόρου άνθρακα θα το περάσω γρήγορα, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Ας μην ξεχνούμε και άλλες πηγές, το φυσικό αέριο, που δεν αναφέρεται πάρα πολύ συχνά. Θα πρέπει να στηρίζουμε περισσότερο και την έρευνα. Να μην επενδύονται χρήματα σε λιγότερο χρήσιμες μεθόδους. Το θέμα της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα. Έχουν δοθεί πολλά κονδύλια σε προγράμματα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, αλλά δεν έχουμε αρκετά επιστημονικά τεκμήρια ότι σε μεγάλη κλίμακα είναι λειτουργικό αυτό το σύστημα και αποδοτικό. Και ότι μπορεί να δεσμεύσει και να αποθηκεύσει μεγάλες ποσότητες άνθρακα. Ε, άλλο που είναι και πολύ δαπανηρό αυτό το σύστημα. Οπότε αυτά τα κονδύλια, αντί να τα χορηγούμε σε τέτοιου είδους ε, αναποτελεσματικά μέσα, γιατί να μην τα επενδύσουμε σε άλλες τεχνολογίες, σαν αιμογεννήτριες για παράδειγμα, που έχουν πολύ πιο άμεσα αποτελέσματα και δεν χρειάζεται να περιμένουμε 15-20 χρόνια και να είναι και αβέβαια η έκβασή τους. Επίσης, ε, σκόπιμο θα ήταν να εξετάσουμε το θέμα και πέραν των οικονομικών κριτηρίων. Έχετε για το 2007 κάποια στοιχεία και οικονομικά και έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και βλέπετε ότι οι περισσότερες πολιτικές στήριξης ακολουθούν την πορεία των χρημάτων. Όπου βρίσκονται τα χρήματα εκεί κατευθύνονται και άλλα κονδύλια. Για παράδειγμα οικονομίες άνθρακα. Γιατί λοιπόν να μην διερευνηθούν και άλλες μέθοδοι Ίσως η χρηματοδότηση, η συγχρηματοδότηση θα είναι μια λύση. Γιατί όταν ζητάτε συγχρηματοδότηση, συνήθως ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που συμμετέχει. Αλλά μερικές φορές μένουν εκμετάλλευτες κάποιες τεχνολογίες. Για παράδειγμα, έξυπνοι μετρητέ, ε, αποθήκευση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευφυή δίκτυα. Αυτά δεν αναφέρονται παρκώς σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των εταιριών. Και δύο λεπτά στο τελευταίο ομιλητή. Το τελευταίο στοιχείο που θα θέλαμε να σας αναφέρουμε, το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην θεωρία, θα πίστευε κανείς ενδεχομένως ότι ότι όλα αυτά τα θέματα της αποκεντρωμένης ενέργειας και της ανταπόκρισης στη συζήτηση θα έπρεπε να είναι φιλικά προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί μειώνει το κόστος ενέργειας, και καταστά τις λιγότερο εξαρτημένες από τις τιμές των καυσίμων και ενδεχομένως να αποτελέσουν και περαιτέρω πηγή εσόδων. Γιατί όταν χρησιμοποιεί κανείς, ε, όταν παράγει κανείς ηλιακή ενέργεια μπορεί να την πουλήσει στο δίκτυο το δημόσιο. Αυτό θεωρητικά. Στην πράξη όμως προκύπτουν μια σειρά προβλημάτων. Καταρχάς η αποκεντρωμένη ενέργεια επιβαρύνεται από ένα μεγάλο αρχικό κόστος, κεφάλαιο. Γιατί ο χρόνος απόσβασης είναι πολύ μεγάλος. Ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πολύ πιο βραχή ορίζοντα. Επίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συχνά δεν γνωρίζουν, δεν γνωρίζουν τι δυναμικό εξοικονόμηση ενέργειας υπάρχει ή ότι μπορούν για παράδειγμα να πουλήσουν στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης την ενέργεια που παράγουν. Υπάρχει συχνά ένα τεράστιο κενό προς την εξειδίκευση και γνώση. Και μόνο οι μεγάλες ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν κάποιον ειδικό για τέτοια θέματα ενέργειας. Άρα, προτείνουμε να γίνει πολύ πιο έντονη και εντατική ενημέρωση, να υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία όπως το Energy Tool Και να μην υπάρχουν ε, εμπόδια. σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να περάσουμε τώρα στα συμπεράσματα. Στην τελευταία διαφάνεια αναφέρουμε τα βασικά πορίσματα της ε, έρευνάς μας. Καταρχάς θα συστήναμε τη βελτίωση των διασυνδέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τρίτο ενεργειακό πακέτο σαφέστατα αποτελεί ένα καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να ε, παρακολουθείτε καλύτερα και να εφαρμοστεί. Έχουμε την εντύπωση ότι το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πολύ φιλικό στα μεγάλα, μεγάλης κλίμακας ε, project, αλλά όχι για τα μικρά. Θα θέλαμε λοιπόν αυτή η πτυχή να διορθωθεί. Γνωρίζουμε φυσικά ότι υπάρχουν φορολογικά ζητήματα τα οποία είναι ευαίσθητο θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόλα αυτά ε, προτείνουμε ε, φόρο για τον άνθρακα και μία πανευρωπαϊκή κλίμακα για την τιμή του ΦΙΤ. Επίσης θα θέλαμε να προσαρμοστεί το πλαίσιο υποστήριξης ε, έρευνας και τέλος να εξαλευτούν τα εμπόδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί πραγματικά το δυναμικό είναι τεράστιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες αυτές που μας δώσατε. Ο συνάδελφος Γκλάντας έτσι το λόγο. Τελευταίος των Μαϊκανών. Σας δίνω το λόγο λοιπόν. Δεν θα είμαι ο τελευταίος που θα πάρω το λόγο, είμαι βέβαιος, αλλά να ευχαριστήσω για την παρουσίαση τη μελέτη. Έχουν ε, κάποια ερωτήματα, όχι ιδιαίτερα για τα απορίσματα τη μελέτη, αλλά για το μέλλον. Έγιναν διάφορες συζητήσει σε ό,τι αφορά το ενεργειακό πακέτο για το μέλλον, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ιστορική αγορά. Στο μέλλον θα υπάρχουν και θα χρειάζονται μεγάλες ε, δίωδοι από τον βορρά στον νότο. Για παράδειγμα, αν δεν ε, έχουμε αέρα στον νότο, θα έχουμε στον βορρά. Ή για παράδειγμα, φωτοβολταϊκά στον νότο και αντίστροφα. Χρειαζόμαστε λοιπόν τέτοιες, τέτοιους ε, αγωγούς. Αυτούς τους αγωγούς ποιος θα τους διαχειρίζεται και ποιος θα τους χρηματοδοτήσει. Στη Γερμανία γίνεται μία συζήτηση για την αποζημίωση, την αμοιβή τροφοδότησης. Όλα καλά και ωραία, αλλά υπάρχουν προβλήματα. Για παράδειγμα, όταν χρειάζονται εγγυήσεις τιμών για, με βάθος 20 ετίας σε περίπτωση φωτοβολταϊκών. Και φυσικά αυτά περιπλέκονται περαιτέρω σε παρευρωπαϊκό επίπεδο για την αποκέντρωση. Μου είχαν πει πριν από κάποια χρόνια ότι το μέλλον της παραγωγής της ενέργειας θα είναι όπως το διαδίκτυο. Θα υπάρχουν πάρα πολλοί μικροί παραγωγοί. Γιατί να σας ρωτήσω όμως το εξής. Πώς θα διαχειριστούμε και θα καθοδηγήσουμε αυτά τα μικρά, αυτές τις μικρούς παραγωγούς χωρίς να ρισκάρουμε την σταθερότητα του δικτύου. Γιατί χρειάζεται πάνω απ' όλα ασφάλεια. Χρειάζονται ασφάλεια καθοδήγηση των δικτύων αυτών και υπάρχει λοιπόν ένα όριο σε αυτή την αποκέντρωση και αυτό με απασχολεί ειλικρινά. Και μιλάμε για τους μεγάλους αγωγούς ε, ρεύματος, φωτοβολταϊκά, στο, στη Νότια Ευρώπη, στη Βόρεια Αφρική ενδεχομένως. Έστω ότι γίνεται αυτό και θέλουμε ευρωπαϊκή υποστήριξη θα χρειαστεί συνάντηση των κρατών μελών και να αποφασιστεί ένα ενεργειακό μείγμα και θα είναι πραγματικά πολύ ε, έντονη συζήτηση για τα smart grids, για τα FEE ε, δίκτυα, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά άκουσα πρόσφατα πόσα νοικοκυριά θα μπορούσαν να εφαρμόσουν το σύστημα αυτό και πόσο αποδεκτό θα ήταν ένα σύστημα. Για παράδειγμα, να μην βάζει κανείς πλυντήριο κάποια ορισμένη ώρα. Δεν ξέρω αν όλοι θα συμφωνούσαν. Το ψυγείο το καταλαβαίνω πιο εύκολα. Έχει καλή μόνος και θα μπορούσε να μείνει κρύο. Αλλά αυτές οι εξοικονομήσεις ενέργειας μέσω των ε, εφιών δικτύων και των εφιών δικτών, μέχρι που μπορούν να φτάσουν. Γιατί πώς θα καθοριστούν και οι εμπορικές τιμές, ε, πώς θα ξέρουμε την κατανάλωση, πώς θα ξέρουμε πόσο αέρα θα φυσήξει και πόσο, πόσο μεγάλη θα είναι η παραγωγή. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να συζητηθούν. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος, αυτά τα ερωτήματα τα απευθύνω και προς τους ειδικού μας. Oh, συγγνώμη. Η κυρία Ματία ζήτησε το λόγο για να θέσει και αυτή η ερωτήση. Συγγνώμη, δεν σα πρόσεξα. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονε για την παρουσίαση της μελέτης για ένα τόσο σημαντικό θέμα για την Επιτροπή μας. Έχω μία ερώτηση για ένα σημείο που αναφέρατε τη βελτίωση των διασυνδέσεων ενεργειακής μετάδοσης. Αυτό είναι σημαντικό σημείο για τρεις λόγους. Καταρχήν γνωρίζουμε ότι αυτή η βελτίωση των διασυνδέσεων είναι σημαντική γιατί σε επίπεδο διασυνδέσεων είναι που έχουμε μεγάλη απώλεια ενέργειας. Έχετε άλλες πιο συγκεκριμένες προτάσεις από αυτές που αναφέρονται στα συμπεράσματά σας γιατί αν υπάρχουν θα ήθελα να τις μάθω. Όταν μιλούμε για ανανεώσιμες ενέργειες, γνωρίζουμε ότι πολλά κράτη-μέλη δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα με τους προκαθαρισμένους στόχους και το ποσοστό ανανεώσιμης ενέργειας ενώ άλλες χώρες μπορεί με να παράγουν το ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως οφείλονται, αλλά δεν μπορούν να τη διοχετεύσουν μετά. Και αυτό είναι πραγματικά κρίμα. Και τελευταίο θέμα που σχετίζεται με το προηγούμενο. Είναι ότι εμείς εξετάζουμε τα συστήματα παραγωγής σε ευρωπαϊκή κλίμακα και μιλούμε μεν για την αποκέντρωση, αλλά φαίνεται να ξεχνούμε κάτι που επίσης είναι πολύ σημαντικό, της παραγωγή σε μικρή κλίμακα. Γιατί μιλούμε για παραγωγή μεγάλης κλίμακας και καλώς κάνουμε και για την αποκέντρωση, αλλά τι γίνεται με την παραγωγή μικρής κλίμακας. Νομίζω ότι και εκεί θα χρειαζόμασταν μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση της ε, παραγωγής σε μικρή κλίμακα, μικροπαραγωγής. Έχετε το λόγο. Να προσπαθήσω να απαντήσω. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. I, guess the, first question, real big... Η, η πρώτη μεγάλη ερώτηση ήταν το πώς θα τα χρηματοδοτήσουμε όλα αυτά, γιατί πολλά φυσικά προτείνω τα οποία όμως κοστίζουν χρήματα. Και κάποιος τελικά θα πρέπει να πληρώσει το λογαριασμό και κάποιος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο και για την διαχείριση των συστημάτων αυτών. Να αναφέρω στο σημείο αυτό ότι τα ενεργειακά συστήματα θα πρέπει να, έχουν, να υπάρξουν επενδύσει προ τα ενεργειακά συστήματα ούτως ή άλλως τα επόμενα χρόνια, γιατί θα αυξηθεί η ζήτηση. Κατά 2% εκτιμάται ανά χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά από κάπου που θα πρέπει να έχουμε ενέργεια, να προέλθει αυτή η ενέργεια και κάπως θα πρέπει να τη χειριστούμε την ενέργεια αυτή. Άρα φαντάζομαι ότι το μεγάλο ερώτημα δεν είναι ποιος θα τα πληρώσει αυτά και πώς. Το μεγάλο ερώτημα είναι πού θέλουμε να ξοδεύσουμε τα χρήματά μας, γιατί κάπου θα πρέπει να αφιερώσουμε τους πόρους αυτούς και κάποιος θα πρέπει να διαχειριστεί τα συστήματα αυτά. Άρα το ερώτημα δεν είναι ουσιαστικά πραγματικό ερώτημα. Ασφαλώς και θα κοστίσουν χρήματα. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε νέο σύστημα για την ενέργεια, οποιοδήποτε ενεργειακό μοντέλο θα κοστίσει χρήματα. Το πλεονέκτημα του αν βασιστούμε σε ένα σύστημα ε, ανανεώσιμων είναι ότι θα είναι καλύτερο από το σύστημα που έχουμε σήμερα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και τις, ε, τους στόχους που έχουμε θέσει για το περιβάλλον. Αν θέλουμε να συζητήσουμε θέματα κόστους, δεν είμαι πεπισμένος ότι το σύστημα που βασίζεται στις ανεώσιμες και στις αποκεντρωμένα συστήματα ενέργειας είναι πιο ακριβό. Το αντίθετο, ίσως. Έχουμε και κάποιες ε, λεπτομέρειες στην έκθεση για το κόστος των διαφόρων τεχνολογιών και το βασικό επιχείρημα είναι ότι οι ανανεώσιμες είναι, γίνονται όλο και πιο φτηνές, ενώ οι τεχνολογίες ορεικτών καυσίμων καθίστανται όλο και πιο ακριβές. Λόγω των αλλαγών της προόδου της τεχνολογίας, οι ανανεώσιμες ενέργειες γίνονται όλο και πιο φθηνές. Άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Μιλάτε για τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Η διασύνδεσή τους θα τα καταστήσει πολύ πιο αποδοτικά σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ρεύματος. Το τελικό κόστος θα είναι πιο μικρό, παρά το γεγονός ότι θα κοστίσει φυσικά η δημιουργία τους. Άρα τελικά πιστεύω ότι πιο πολλά χρήματα θα εξοικονομήσουμε παρά θα ξοδέψουμε. Ποιο θα είναι υπεύθυνο της διαχείρισης. Αυτά είναι βασικά θέματα, μεγάλα προβλήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν, αλλά κάποιοι είναι υπεύθυνοι και σήμερα για τα συστήματα αυτά ενέργεια. Ήδη φαντάζομαι θα διαχειρίζονται και τα μελλοντικά συστήματα. Σίγουρα από κάποιους θα τα διαχειρίζεται. Για την ε, διασύνδεση των δικτύων ε, ενέργειας, συγκεκριμένες προτάσεις τώρα. Δεν έχουμε πολλές περισσότερες συγκεκριμένες προτάσεις παρά από αυτές που συμπεριλαμβάνονται στην μελέτη. Η ανάπτυξη των διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών θεωρώ ότι είναι ουσιώδης σημασία. Άρα Αλλιώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά τα δίκτυα. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη λύση πραγματικά. Προφανώς οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, τα κονδύλια για τις διασυνδέσεις αυτές θα βοηθήσουν να υπάρξουν σχετικά προγράμματα προς την κατεύθυνση αυτή να σας πω ότι δεν ήταν ε, εντολή μας να αναπτύξουμε νέες πολιτικές. Ενδιαφέροντα να απαντήσουν τα ερωτήματα που θέσατε. Επίσης, ρωτήσατε ποια τεχνολογία θα πρέπει να προτιμηθεί. Δεν κατάλαβα ακριβώς γιατί το ρωτάτε αυτό. Γιατί σας απασχολεί αυτό. Αν θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε τι θέλετε να μάθετε, Ασφαλώς κάθε χώρα μπορεί να επιλέξει την τεχνολογία που της ταιριάζει καλύτερα και αυτό φυσικά είναι διαφορετικό ανά χώρα. Πάντα υπάρχουν όμως τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θερμικές αντλίες θερμότητες, ε, για παράδειγμα. Υπάρχουν πάρα πολλές, πολλές μορφές και δυνατότητες για την αξιοποίηση ενεργειακών ανέωσιμων πηγών ενέργειας. Όντω διαφέρουν τα χαρακτηριστικά αυτά από χώρα σε χώρα. Οι πόροι επίση μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα για τη χρηματοδότηση των, των προγραμμάτων αυτών. Συχνά ακούω το επιχείρημα ότι, για παράδειγμα, στην τάδε χώρα δεν υπάρχουν τα κονδύλια για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων. Ε, υπάρχουν όμως πολλοί επενδυτές οι οποίοι θα ήθελαν να επενδύσουν αν υπήρχαν οι κατάλληλε δομέ για επενδύσεις. Πραγματικά είναι πολύ άριθμοι οι επενδυτές. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι οι πόροι αποτελούν αποτρεπτικό εμπόδιο. Αν ε, με την ερώτηση υπονοούσατε την πρόταση για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα FIT, δεν ξέρω. Το πλεονέκτημα του συστήματος FIT γενικότερα είναι, ανακρατός μέλος, ότι μπορεί κανείς να υποστηρίξει τις τεχνολογίες που επιθυμεί με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν χρειάζεται να προτιμηθούν, για παράδειγμα, τεχνολογίες οι οποίες δεν έχουν νόημα σε κάποια κράτη-μέλη. αν θέλουμε τώρα και ένα πανευρωπαϊκό σύστημα FIT πέρα από τα εθνικά συστήματα FIT, το μοναδικό πλεονέκτημα που συνηγορεί υπέρ αυτού είναι να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο τεχνολογιών σε κάθε χώρα για όσους ενδεχομένως θέλουν να αναπτύξουν τις τεχνολογίες αυτές και θέλουν ε, υποστήριξη από ένα πανευρωπαϊκό σύστημα. Ελπίζω έτσι να απάντησα την ερώτησή σας. Gut, ich mich. Ja, bitte. Very, very briefly. Δύο λόγια μόνο. Επανέρχομαι στο θέμα της τιμής των ανανεώσιμων. Κάτι που με εκπλήσει κάθε φορά είναι ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιεί κανείς ανανεώσιμες ενέργειες και επενδύσει αυτές, τόσο πιο φθηνές γίνονται. Ενώ με τα ρηκτά καύσιμα, όσο περισσότερο τα χρησιμοποιεί κανείς, τόσο περισσότερα κρυβαίνουν. Νομίζω ότι και μόνο αυτό είναι επαρκής λόγος για επένδυση σε αποκεντρωμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεύτερο, συναφές με το ερώτημα για τα εφή δίκτυα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγενίασε την εισαγωγή των έξυπνων μετρητών με στόχο 80% των νοικοκυριών μέχρι το 2020 να έχουν έξι προσμετρητές. Πολύ καλό βήμα νομίζω. Για να βελτιστοποιήσουμε την κατανάλωση ενέργειας και σε επίπεδο νοικοκυριών και καταναλωτή. Βέβαια δεν θα είναι χρήσιμο το μέτρο αν ταυτόχρονα δεν ε, ε, εισαχθούν, δεν θεσπιστούν κειμενόμενες τιμές ηλεκτρισμού για τον καταναλωτή. Γιατί τέτοιες κειμενόμενες τιμές ηλεκτρισμού θα επιτρέψουν ε, real-time επικοινωνία μεταξύ του καταναλωτή και του διαχειριστή του δικτύου και πραγματικά βελτιστοποίηση σε πραγματικό χρόνο της ενεργειακής κατανάλωσης. Ευχαριστώ. Στα κανείς άλλο το λόγο, λέει ο Πρόεδρος να ευχηθώ καλό ταξίδι στους συναδέλφους, να ευχαριστήσω τους εμπρεγνώμονες, τους υπαλλήλους μας που ήταν μαζί μας και καλή επιστροφή σας εύχομαι στα σπίτια σας.